θέλει η κυρία Πρόης ε, να συμμετάσχει στην Ισομερή Συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θέση της κυρίας Γκέπχαρτ. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις? Όχι. Η Επιτροπή Ήμικο ενέκρινε μία σύσταση